Λοιπόν, καθίστε παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε καθυστερήσει ήδη ένα τέταρτο. Ελπίζω να θυμηθήκατε να φέρετε τι ηλεκτρονικέ σα κάρτε για τι ψηφοφορίε. Αν όχι, πηγαίνετε να τι φέρετε, γιατί έχουμε πολύπλοκε ψηφοφορίε να διεκπαιρεώσουμε. Λοιπόν, Καταρχάς ε, κάποιος με ρωτάει αν θα μας σερβίρουν καφέ και τσάι. Λοιπόν, μετά τις ψηφοφορίες είναι η απάντηση, όχι όσο θα ψηφίζουμε. Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθατε όλες και όλοι. Ξεκινούμε την συνεδρίασή μας με το πρώτο σημείο έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης. Έχετε μήπως αντιρρήσεις ή κάποιο σχόλιο. Όχι, επομένως η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Επόμενο σημείο, έχετε λάβει τα πρακτικά της συνεδρίασης της 29ης και 30ης Αυγούστου του 2011. Αν έχετε αντιρρήσεις παρακαλώ να ενημερώσετε τη γραμματεία πριν από το τέλος ε, της ε, σημερινής μας συνεδρίασης. Αλλιώς θα εγκριθούν τα εν λόγω πρακτικά. Έχουμε ένα λεπτό για τις ερωτήσεις ε, προς την Κομισιόν. Δεν λάβαμε όμως κάποια ερώτηση και περνάμε στο επόμενο θέμα ανακοίνωση τη Πρόεδρου. Δεν υπάρχουν ανακοινώσει από πλευρά μου και επομένως μπορώ να περάσω στο επόμενο σημείο. Έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια ανακοίνωση. Ναι. Ο κύριος Ντομέν Κορόσα, έχετε το πολύ δύο λεπτά. Ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ξέρω ότι έχετε ψηφοφορίες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ε, για την ε, ανάπτυξη. Το Νοέμβριο θα διεξαχθεί και θέλαμε να συζητήσουμε τις ανακοινώσεις ε, που σας παρουσίασε σε αδρές γραμμές η συνάδελφός μου στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης. Νομίζω ότι με τα κράτη-μέλη θα μπορούσαμε να έχουμε μία συζήτηση γενικού προσανατολισμού για το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τον αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ανάπτυξης, καθώς επίσης και το μέλλον της δημοσιονομικής υποστήριξης. Κάτι άλλο που θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον για την Επιτροπή σας είναι ότι μέχρι τα τέλη του έτους η Κομισιόν θα δημοσιεύσει κατά πάσα πιθανότητα την έκθεσή της για την συνοχή, τη συνεκτικότητα των ε, πολιτικών ένα θέμα που περνούσε λίγο παρατήρητο τα προηγούμενα χρόνια και ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε μεγαλύτερη προβολή ε, και να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με την έκθεση για όσες πτυχές ενδιαφέρουν την Επιτροπή Ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περάσουμε στην ε, ψηφοφορία με βάση τον κατάλογο ψηφοφοριών. Λοιπόν, τις κάρτες σας παρακαλώ όλοι και εγώ πρέπει να βγάλω τη δική μου μισό λεπτό. Alors, Merci. Alors, est-ce que vous avez tous votre carte? Λοιπόν, έχετε όλοι τις κάρτες σας. 3, 2, 1. Ωραία. Alors, nous allons passer au premier vote. Λοιπόν, ξεκινάμε με την ψηφοφορία. Όχι. Α, ναι, πρέπει να κάνουμε μια δοκιμή πρώτα. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία, δοκιμαστική. Δοκιμή κάνουμε, κύριε Μπέρμαν, για να δούμε αν λειτουργούν οι κάρτες. Λοιπόν, πέρα της ψηφοφορίας, για να δω πόσους βουλευτές έχουμε. Λείπουν βουλευτές. Έχετε ψηφίσει όλοι. Να ξαναδοκιμάσουμε παρακαλώ. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Περιμένω να τοποθετήσετε όλοι τις κάρτες στο μηχάνημα. Λοιπόν, πέρασε τη δοκιμαστική ψηφοφορία. Νομίζω τώρα είμαστε εντάξει. Ωραία.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 Λοιπόν, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη βιομάζα και ο αντίκτυπός της στην ανάπτυξη. Τροπολογία 1. Το κάνουμε χρονικά. Όχι. Αδιανατάσσω στις χειρός. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τελική ψηφοφορία για την προφορική ερώτηση. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Alors, Λοιπόν, τώρα η ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, το ψήφισμα. Είναι λίγο πολύπλοκα σήμερα τα πράγματα, λέει Πρόεδρος. Λοιπόν, έγκριση πρότασης ψηφίσματος, τροπολογία 27, ψήφι υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 29 σε δύο τμήματα υπέρ, κατά, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 29. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, ηλεκτρονική ψηφοφορία μάλλον καλύτερα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Λοιπόν, τροπολογία 30 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, διανατάσσω χειρό παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πρώτη προφορική τροπολογία ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα δεν έχω καταλάβει και μπερμάνε ψηφίστε υπέρ ή κατά. Λοιπόν, τροπολογία 32. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία όχι, όχι καταπίπτει. Επομένως πάμε στην τροπολογία 33, όχι. Και αυτή έχει καταπέσει. Άρα περνάμε στην προφορική τροπολογία 3, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 34, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 35, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 36, 36 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 σε δύο τμήματα υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Προφορική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 κατά πι, τροπολογία 39 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Κύριε Σαρτζεντίνη, απορρίπτεται κύριε Σαρτζεντίνη, θέλετε το λόγο. Η κάρτα μου δεν έχει έρθει ακόμα και ήθελα να ψηφίσω υπέρ και εγώ. Και η κυρία Κέλλερ. Απλά σα το αναφέρω. Okay. Εντάξει, λοιπόν, τροπολογία 40 υπέρ. Α, ξέχασα την 39, λέει πρόεδρος, με συγχωρείτε. Μα αυτό που δεν ψηφίσαμε τώρα. Και δεν έγινε δεκτό. Ωραία, λοιπόν, άρα πάμε στην τροπολογία 40. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική 5 ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 41. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ. Κατά. Αποχές θα το ελέγξουμε. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 43. Πέρας. Εγκρίνεται, αλλά... Ξεχάσατε τις κάρτες, ε, εντάξει, μας κάνετε να δουλεύουμε 10 φορές παραπάνω με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Μα ε, τι γίνεται. Κανονικά δεν μπορώ να δεχθώ ε, ψήφους που γίνονται διαλαντά στους χειρός όταν έχουμε όμως ψηφίσει εμείς ηλεκτρονικά. Τρία χρόνια το κάνουμε αυτό. Ε, κάποια στιγμή, τι να σας πω, δεν είναι και τόσο πολύπλοκο να σκεφτείτε να φέρετε τις κάρτες σας. Κύριε Κέλλερ, πείτε μας ποιοι δεν έχουν κάρτες τώρα. Εσείς ε, σας τη φέραν τη δική σας. Λοιπόν, κατεξαίρεση γίνεται αυτό. κατεξαίρεση σε διάφορες περιπτώσεις άλλοι έχουν χάσει τις κάρτες τους και ποτέ δεν έχει αποτελέσει αυτό πρόβλημα. Ναι, φυσικά είναι πρόβλημα που δεν έχω τώρα την κάρτα μου. Πολύ λυπάμαι, δεν είναι όμως η πρώτη φορά. really also... Και επίσης υποτίθεται ότι θα ξεκινούσαμε στις 10. Ε, λυπάμαι που άργησα, αλλά δεν θα μπορούσαμε να το κοιτάξουμε αυτό. Λυπάμαι για την κάρτα μου, αλλά δεν είμαι και η πρώτη που έχει ξεχάσει την κάρτα της. Λοιπόν, πράγματι συχνά το δεχόμαστε, αλλά ε, κάποια στιγμή σε κάποιες πολιτικές ομάδες έχουν υπάρξει καταχρήσεις. Και σε κάποιες περιπτώσεις ε, δεν δεχόμαστε να ψηφίσουμε χωρίς κάρτες γιατί χάνουμε τον μπούσιλο ορισμένε φορές. Λοιπόν, υπάρχουν κείμενα και δεν μπορούμε να δεχόμαστε ψήφους ε, διανατάσσεως χειρός όταν έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κάποιες εξαιρέσεις κάνουμε, αλλά αν δεν είμαστε αυστηροί ε, θα έχουμε χάος για τρία χρόνια. Γιατί κάποιες φορές χρειάζεται να τα υπολογίζουμε από την αρχή όλα και να κάνουμε υποσημειώσεις και τα λοιπά. Είναι θέμα λογικής και είναι και ζήτημα σεβασμού. Όταν έχουμε ψηφοφορίες φέρνουμε τις κάρτες μας. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, κατ' εξαίρεση, αλλά όχι από εδώ και πέρα αν είμαι εγώ πρόεδρος. Είναι τελευταία φορά που κάνω εξαιρέσεις. Πρέπει να πειθαρχήσουμε λίγο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κασμάρ και μετά θα περάσουμε σε ψηφοφορία. Ο κύριος Κάσμαρ. κύριος Κασμάρ. Ο κύριος Κάσμαρ. Ευχαριστώ, ε, πρόεδρε. καταλαβαίνουμε και δεχόμαστε τη θέση σας, αλλά έχει δίκιο και συνάδελφος σε κάποιες άλλες επιτροπές και σε αυτή την επιτροπή δεν τον εφαρμόζαμε τον κανόνα αυτό που θα έπρεπε, όπως είπατε, αλλά θεωρώ ότι είναι δίκαιο όχι επειδή δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές και σεβαστές οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Όχι, πρέπει να γίνονται και αυτό διευκολύνει και τη δική σας τη δουλειά και τη δουλειά της Επιτροπής. Αλλά κοιτώντα τι γινόταν μέχρι τώρα, γινόταν ε, καταγραφή της ψηφοφορίας και της ψήφου των βουλευτών ακόμα και χωρίς κάρτα. Λοιπόν, οι ψηφοφορίε γίνονται διανατάσσεω τη χειρό και όταν υπάρχει αμφιβολία ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρα εκ των προτέρων δεν μπορούμε να γνωρίσουμε αν θα υπάρξει κάποια αμφιβολία για κάποια ψηφοφορία. Λοιπόν, τώρα θα χάσουμε ένα τέταρτο συζητώντα το θέμα αυτό. Εγώ αυτό που προτείνω απλά είναι να ψηφίσουμε. Λοιπόν, θα δεχθούμε ε, και κάποιου που ψηφίζουν χωρί κάρτα ή όχι. Κύριε Γκέρεν, θα είσαι το τελευταίο που θα λάβει το λόγο, αλλά αρχίζω να εκνευρίζομαι. Κύριε Γκέρεν. Τόσο πολύ μας φοβήσατε που βρήκε και την κάρτα της η κυρία Κέλλερ. Ωραία. Τέλεια λέει η πρόεδρος. Χαίρομαι όλους ιδιαιτέρως. Από εδώ και πέρα δεν θα δεχθώ ψήφο χωρίς κάρτα. Εάν βέβαια ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αν δεν εφαρμόζουμε τους κανόνες κάποια στιγμή μετά από κάποια χρόνια δεν θα υπάρχει καν κανένας κανόνας και θα υπάρχει χάος. Αυτό δεν είναι λογικό. Επειδή κάποιοι δεν τηρούν τους κανόνες, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να του εφαρμόζει κανεί. Λοιπόν, κατ' εξαίρεση ξαναρχίζουμε αφού έχουμε ε, την κάρτα και της κυρία Κέλλερ. 43 τροπολογία ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ, κατά, ηλεκτρονική ψηφοφορία 46 τροπολογία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 47 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 49. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Α, όχι. Έχει αποσυρθεί. Τι ψηφίζουμε τώρα. Χωριστή ψηφοφορία για την παράρφο 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι η χωριστή ψηφοφορία επί της παραγράφου 10. Αρχικής παραγράφου 10. Εντάξει. Απορρίπτεται. Λοιπόν, ιδεολογικές σκέψεις. Recital. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να το ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Βλέπετε η ισοψηφία και απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 7 πρώτο τμήμα τι θέλετε να ελέγξουμε ελέγχουμε την 6 την 6 τροπολογία πέρας το ίδιο 10 όλα απορρίπτεται κι αυτή είχατε δίκιο Λοιπόν, τροπολογία 7, δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, υπάρχει και τρίτο τμήμα, συγγνώμη, δεν το είχα δει. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε όμως. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 8. Πέρας. Πράγματι απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ του πρώτου τμήματος παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, προφορική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 14 κατά πίπτη. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 16 υπέρ, κατά. Ας το ελέγξουμε καλύτερα, νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε. Τροπολογία 16 ηλεκτρονικά, παρακαλώ περαση ψηφοφοριας ψηφοφορίας. στο ψηφια ισοψηφία 10-10, επομένως, τι να πω, συνέχεια αυτό γίνεται, απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, όχι, καταπίπτει. 19 υπέρ, κατά, ας το ελέγξουμε. Τροπολογία 19 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά. Ας το ελέγξουμε. Τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά. Ελέγχουμε τροπολογία 24, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Χωριστή ψηφοφορία λοιπόν για το και λατινικό. Ποιοι είναι υπέρ. Α, όχι. Κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Τροπολογία 25. Κάποιος λείπει. Πέρας ψηφοφορίας. Να περιμένουμε λίγο. Αν έχετε την κάρτα σας. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι θα απορριφθεί ψηφία νομίζω ότι υπάρχει, αλλά λοιπόν, ας περιμένουμε. Ας περιμένουμε. Εντάξει, ψηφίσατε κι εσείς, ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν. Χάρη στην κυρία Ντεκεζέρ και θα πρέπει να την ευχαριστήσετε. Λοιπόν, τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται Χωριστή ψηφοφορία. Όχι, καταπίπτει. Καταπίπτει. On vote les citations. Amendement numéro 1. Λοιπόν, ψηφίζουμε τις ε, αναφορές στα citations. Τροπολογία να δεχτεί. Δεύτερη, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα Τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Le vote est clos. Adopté. Εγκρίνεται. Κυρία Πρόεδρε, μπορούμε να κάνουμε την πρώτη σελίδα μαζικά, ίσως. Για την έκθεση Κασμάρεκ, ε, η πρώτη σελίδα, όπως φαίνεται, δεν γίνεται να ψηφίσουμε μαζικά. Θα το κάνουμε για μερικά τμήματα, αλλά όχι για όλη τη σελίδα, γιατί όπως βλέπω υπάρχουν διαφορετικές ψήφοι. Ah, Oui. bon, allez, euh, on, on continue. Συνεχίζουμε λοιπόν, προτείνουμε λοιπόν μαζί την τροπολογία 7 και 8 υπέρ κατά αποχή. Εγκρίνεται 9 κατά. Νομίζω ότι είναι υπέρ, αλλά ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία μπορούμε να κάνουμε μαζί. Πιστεύω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε μέχρι το τέλος. Μέχρι την 25 στο ΕΛ και είμαστε υπέρ. Αν δεν υπάρχει άλλη διαφορά άποψη, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες. Εγώ είχα ένα πλήν, συνεπώς υπήρχε κάποιο λάθος. Κύριε Κάσμαν, θέλατε το λόγο. Μισό λεπτό κύριος Κάσμαν, έχει το λόγο. Ναι, έτσι είναι. Μέχρι το 26, επειδή είναι ξεχωριστή η ψηφοφορία, μέχρι και το 25. Και το 25 μαζί δηλαδή. Ψηφίζουμε λοιπόν σε μπλοκ μέχρι το 25. Ε, όχι, συμπεριλαμβάνεται λάθο το 24. Λοιπόν, συνεχίζουμε, διότι εδώ δεν βρίσκουμε άκρη. Λοιπόν, που ήμασταν στην 10 έως την 15. Υπέρ, κατά, αποχή, εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ψηφίσουμε μαζικά από τη 17 έως την 24 έως και την 24 ναι υπέρ κατά αποχή εγκρίνεται τροπολογία 25 έως και 27 όχι λάθος 25 μόνο υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά. Οι εγκρίνεται 27 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, για τα εκτιμώντας όλα μαζί υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν και τα citations μαζί υπέρ κατά εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική, άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. με ομοφωνία. Η έκθεση του κυρίου Πρέντα. Τροπολογία 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Πάει πολύ γρήγορα. Μόλις με έκαναν παρατήρηση ότι πηγαίνω πολύ γρήγορα. Κυρία... Πρόεδρε, να πω ότι ε, από την Επιτροπή εκ μέρους τη της Επιτροπής ότι είστε η πιο αποτελεσματική και γρήγορη πρόεδρος που είχαμε ποτέ. Ε. Λοιπόν. Merci beaucoup, Monsieur Cashman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάσμαν. Πού είμαστε τώρα, χάθηκα πάλι. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 22 σε δύο κομμάτια το πρώτο μέρος πρώτο μέρος συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μην ε, μου πλέκετε το εγκόμιο γιατί μετά τα χάνω δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική ε, α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Είμαστε λοιπόν στην τροπολογία 28, υπερκατά, κατά, αποχές απορρίπτεται, 29 υπέρ, κατά, ε, θα ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται, τέλος ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Δεν βλέπω πολύ καλά, γι' αυτό κοιτάω σε εσά. Ε, τροπολογία 30. Σε δύο μέρη, πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές. Ελέγχουμε με ηλεκτρονική άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Σε δύο μέρη πρώτο μέρος. Σε δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 ε, που καταπίπτει 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ ακαταπίπτει και το 36 38 το 36. Η τροπολογία 36. Συγγνώμη. Νομίζω ότι αν θυμάμαι καλά, η 34 δεν ε, κατέπεσε. Α, κατέπεσε. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε 35. Απορρίφθηκε η 34 και άρα Α, συγγνώμη. Συγγνώμη, Πρόεδρε, έχετε απόλυτο δίκιο γιατί δεν κάθομαι να σα ακούσω καλύτερα. 35 Το 35 καταπίπτει αν η προφορική 1 γίνει, εγκριθεί. Συνεπώ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θέλετε να με μπερδέψετε, κύριε Κάσμαν. Συνήθω είναι ο κύριο Γκέρεν και τώρα εσεί μου κάνετε κόλπα. Ε, τροπολογία 36. Συγγνώμη. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 σε δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεν είμαι σίγουρη θα το ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται για το πρώτο μέρος πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται είδατε έκανα λάθος δεύτερο μέρος υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39 ε, ε, καταπίπτει. Συμβιβαστική σε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 40 καταπίπτει. Συμβιβαστική B υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει λοιπόν και αυτό. Το 42 επίσης καταπίπτει. Τροπολογία 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 43 43, 44, 45 καταπίπτουν. Φτάνουμε στην προφορική τροπολογία 3. Σε δύο μέρη, ποιος είναι υπέρ του πρώτου μέρους, κατά, αποχές, δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, δεν είμαστε σίγουροι. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το δεύτερο μέρος. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 47 καταπίπτει. 48 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος του 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 54 υπέρ ε, καταπίπτει. 55 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 καταπίπτει 57 υπέρ ε, θα ψηφίσουμε μαζί για τις τροπολογίες 57 και 58 πρόκειται για τις ίδιες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σε 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 καταπίπτει συμβεβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 καταπίπτει 65 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε για την 65 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 καταπίπτει. 68 και 69 καταπίπτουν. Τροπολογία 70 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε για τα εκτιμώντας. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 7 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές ε, θα ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 7 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 κατά ε, καταπίπτει τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 5 δεν είναι αποδεκτή. Συνεχίζουμε λοιπόν με τροπολογία 13. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 14 η, ε, ο κύριος Μπέρμαν κάνει απεργία. 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λέω ότι κάνετε απεργία επειδή δεν βλέπω να σηκώνετε το χέρι σας. τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 17 σε δύο μέρη υπέρ του πρώτου μέρους κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 18, 19 υπέρ 18 συγγνώμη έκανα λάθος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με τα... στις αιτιολογικές αναφορές λοιπόν τροπολογία υπέρ κατά εποχές εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική άρχιτη ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, ομοφωνία εγκρίνεται. Alors, je laisse courir la troisième personne. Alors, le rapport de Monsieur Neuser. Λοιπόν, έκθεση Νόιζερ τώρα. Έτοιμοι όλοι. Λοιπόν, τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. 2 και 3. 2 και 3 υπέρ. Υπάρχει ένα πρόβλημα πουθενά. Όχι. Να ξαναρχίσω. Τροπολογία 2 και 3 μαζί. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία για τις τροπολογίες 2 και 3. Πέρασε. Απορρίπτονται. Τοπολογιά 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 και 7 υπέρ. Κατά ελέγχουμε. Τις τροπολογίες 6 και 7 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνονται.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 Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε. Τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ε, ηλεκτρονικό τρόπο. Ομόφωνα λοιπόν δεκτή. Και θα ψηφίσουμε τώρα την έξω κύριο Γκέρενς. Έτοιμοι. Λοιπόν, τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά, ελέγχουμε, άρχεται η ψηφοφορία για τροπολογία 2. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και θα περάσουμε στην έκθεση Σαρτζεντίνη. Amendement numéro 1. Απολογία 1. Υπέρ. Μιλάμε την έκθεση της κυρίας Σαρτζεντίνη. Νομοδότηση. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, έλεγχος με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται, πέρας, ψηφο... πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, δεν σηκώσατε χέρια. Ξεκινάμε ξανά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, τροπολογία, προφορική 1, αρχή ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, πέρας ψηφοφορίας, ε, ε, εγκρίνεται, τροπολογία 2, καταπίπτει. 4, Ποιος είναι υπέρ, καταπίπτει και η 4 επειδή η 1 εγκρίθηκε. Α, όχι, η, η τροπολογία 1 απορρίφθηκε. Συνεπώς ψηφίζουμε για το 4. Είμαστε σύμφωνοι. Κύριε Κάσμαν, δεν συμφωνείτε. Ναι, συμφωνώ. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, Πρέπει να αντιδράτε λίγο καλύτερα γιατί ε, ανακατεύονται όλοι. Λοιπόν, θα πηγαίνω πιο αργά. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 4. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ψηφίζουμε για την 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 τροπολογία 7 σε δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 σε δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές ε, ε απορρίπτεται ε, δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 10 υπέρ α, καταπίπτει 11 ε, και 12 υπέρ, κατά, ελέγχουμε με ηλεκτρονική για την τροπολογία 12, άρχεται η ψηφοφορία, για τις 11 και 12, κλείνει η ψηφοφορία, απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται ε, τροπολογία 15 καταπίπτει. Τροπολογίες 16 και 17 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία 16 και 17 άρχεται η ψηφοφορία. πέρα ψηφοφορία Εγκρίνεται. Συμβεβαστική Β. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτει. Εφόσον 16 και 17 εγκρίθηκαν, συνεπώς καταπίπτει η τροπολογία 18, ζητώ συγγνώμη, και η 19 επίσης. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται τροπολογία 21 υπέρ, κατά ε, αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 23 υπέρ κατά θα ελέγξουμε για την 23 αρχέται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική σε συμβιβαστική C. υπέρ όχι καταπίπτει επειδή εγκρίθηκε η 24 Καταπίπτει λοιπόν. Τροπολογία 25. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 26 υπέρ κατά θα ελέγξουμε είναι πολύ κοντά άρχεται η ψηφοφορία για, για την 26 Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 27 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ, ε, καταπίπτει, λάθος. Ε, τροπολογία 30 επίσης, καταπίπτει. Ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής ντε και η D καταπίπτει. Ah η συμβιβαστική D καταπίπτει επίση, ζητώ συγγνώμη. Τροπολογία 31 επίση καταπίπτει. 32 επίση καταπίπτει. Φτάνουμε λοιπόν στην τροπολογία 33. Ποιο είναι υπέρ, κατά. Θα το ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 33. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την τροπολογία 33. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Α, απορρίπτεται, συγγνώμη. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Περνάμε στην έκθεση της κυρίας Ζολή. Είστε έτοιμοι. Έκθεση της κυρίας Ζολή. Συμβιβαστική 1. Σα προτείνω να ψηφίσουμε από το 1 έω την τροπολογία 2. Και την τροπολογία 2. Ποιο είναι υπέρ από το 1 μέχρι και το 2. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Α, καταπίπτει. 3. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το, από το 6 μέχρι το 9 οι τροπολογίες καταπίπτουν φτάνουμε στη συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 καταπίπτει η τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 1 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 13 καταπίπτει τροπολογία 14 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική άρχεται η ψηφοφορία η τελική ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται η έκθεση ομόφωνα ah Voilà, nous avons ολοκληρώσαμε με τις ψηφοφορίες, μπορούμε να πάρουμε τον καφέ μας. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Ah, merci. Mais j'aimerais bien un café maintenant. Je vous laisse souffler trois minutes puisque vous ne... Αφήνω να πάρετε μια ανάσα για τρία λεπτά επειδή είμαστε πιο νωρίς από ό,τι είχαμε προβλέψει. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο. Είναι εδώ η Επιτροπή. Πότε θα έπρεπε να είναι εδώ στις ε, παρατέταρτο και είναι σχεδόν παραπέντε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Κερδίσαμε λίγο χρόνο και καλό θα ήταν να μην τον χάσουμε. Θα ήταν κρίμα. Γιατί είναι πολύ βεβαρημένη η μερίσια διάταξη. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι περιμένω πέντε λεπτά το πολύ. Όπως ήδη γνωρίζετε, η επόμενη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, παρακαλώ πολύ, θα διεξαχθεί στην Νότια Αφρική, στο Ντέρμπαν, από τις 28 Νοεμβρίου μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2011, μετά από αίτημα της ε, Επιτροπής ΕΝΒΗ, να έχουμε ένα ως το δυνατόν πιο συνεκτικό ψήφισμα μεταξύ των διαφόρων ε, ενδιαφερομένων επιτροπών, οι συντονιστέ Επιτροπή ΔΕΒΕ αποφάσισαν να συμμετάσχουν στο ψήφισμα με ένα σχέδιο κειμένου, το οποίο θα είναι η βάση τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων. Το κείμενο αυτό στη συνέχεια θα τροποποιηθεί και θα εγκριθεί κατά την προσεχή συνεδρίασή μα στι 11 Οκτωβρίου. Θα δώσω καταρχά το λόγο στην Κομισιόν για να μα παρουσιάσει την ανακοίνωση αυτή και εν συνεχεία θα δώσω το λόγο στου βουλευτέ τη Επιτροπή μα. Λοιπόν, ο λόγο στην Επιτροπή. Ποιο θα ήθελε να παρέμβει, παρακαλώ, εκ μέρου τη Κομισιόν. Δεν έχω το όνομα. Παρακαλώ. Εταβού. Euh, euh, Ευχαριστώ πολύ. Ας τα μι... Θα μιλήσω αγγλικά. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο ψηφίσματος. Καλωσορίζουμε το σχέδιο αυτό στην παρούσα μορφή του. Ευχαριστούμε και είμαστε ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο. Ένα σχόλιο να κάνω για τους βασικούς στόχους. Στην δεύτερη παράγραφο των βασικών στόχων αναφέρεται μια έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τις δεσμεύσεις της στη δεύτερη προγραμματική περίοδο. Στην παράγραφο 3 αναγνωρίζεται ότι χρειάζεται συγκριτική πρόοδος για να επιτευχθεί διεθνώς δεσμευτική συμφωνία. Να αναφέρουμε ότι από πλευρά τακτική αν θέλετε, ίσως να μην ήταν και το πιο ε, σόφρον να αναφέρουμε ανοιχτά την προθυμία μας ε, για τέτοια συμφωνία, να συνεχίσουμε αυτές τις συμφωνίες. Νομίζω ότι είναι κάπως υπερβολικό Κατά τα άλλα συμφωνούμε για όλα. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν για το σχέδιο αυτοψηφίσματος όπως έχει στην παρουσιά μορφή του. Okay, Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πάλο Καρίντη και τώρα θα δώσω το λόγο στους βουλευτές. Παρακαλώ, θέλει κάποιος το λόγο? Όχι. Η κυρία Κέλλερ. Ναι, μιλάμε για την έκθεση για τον Τέρβαν, έτσι δεν είναι. Δεν είναι εδώ όμως ο εισηγητής ακόμη. Δεν υπάρχει συγητής, είναι προφορική ερώτηση. Μάλιστα, ωραία. Συγγνώμη. Έχω κάποια σημεία να αναφέρω. Καλωσορίζουμε ασφαλώς την προφορική αυτή ερώτηση. Αγγίζει πολύ σημαντικά θέματα και τα οποία άπτονται και της εργασίας της Επιτροπής Ανάπτυξης γιατί φυσικά όλα αυτά επηρεάζουν και τους δικούς μας τομείς εργασίας. Έχουμε κάποιες προσθήκες, κάποιες τροπολογίες να καταθέσουμε, όπου χρειάζονται διευκρινήσεις. Συμφωνούμε για παράδειγμα πολύ ότι η χρηματοδότηση για το κλίμα θα πρέπει να είναι επιπρόσθετη, αλλά το πρόβλημα με τα επιπρόσθετα κονδύλια αυτά είναι ότι δεν υπάρχει ορισμός για το τι είναι επιπρόσθετο. Άρα, θεωρώ ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα. Άρα σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να υπάρχει και ένας καλός, σωστός, δεσμευτικός ορισμός. Ώστε όταν λέμε, δεσμευτι... όταν λέμε επιπρόσθετα κονδύλια να μην υπάρχει σύγχυση. Επίσης, να αναφερθεί η κόκκινη πρωτοβουλία. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί. γιατί πρόκειται για έναν τρόπο αντιμετώπιση με, φιλικό προ το περιβάλλον τρόπο στην αλλαγή του κλίματο. Επίση, έχουμε το θέμα τη μεταφορά τεχνολογία. Θεωρούμε ότι μπορεί να διδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος μέσω της μεταφοράς της τεχνολογίας, για παράδειγμα στον ενεργειακό κλάδο, σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας ε, και ούτω καθεξής προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και τέλος, στο ίδιο πνεύμα θα θέλαμε το δικαίωμα των ε, αναπτυσσόμενων χωρών να χρησιμοποιήσουν το TRIPS πλήρως, γιατί και αυτό θα επηρεάσει. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι τροπολογίες μας που δεν αντίκειται ουσιαστικά στο πνεύμα της... του σχεδίου, Απλά θεωρούμε ότι θα θέσουν κάποιες επιπρόσθετες ιδέες. Α, και κάτι άλλο. Στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έγινε μια σύντομη συζήτηση για την κλιματική μετανάστευση. Γιατί οι μετανάστες για λόγου κλίματος θα έπρεπε ίσως να συμπεριληφθούν στο σύστημα επικουρικής προστασίας Προτείνουμε λοιπόν και εδώ. Η Επιτροπή Λίμπε είχε δεχτεί μια τέτοια τροπολογία. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα ήταν μια σωστή λύση αυτή για τους μετανάστες για κλιματικούς λόγους, μέχρι ότου υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Monsieur κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με την ε, προηγούμενη ομιλήτρια ότι θα πρέπει να κατατεθούν κάποιες ωφέλιμες τροπολογίες, αλλά φυσικά πάντα στο πνεύμα της ανάπτυξης και σε αυτό το πεδίο εντολής. Θα ήθελα κι εγώ έναν ορισμό των επιπρόσθετων κονδυλίων, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει με μία φωνή στον Τέρμπαν. Όσοι ενδιαφέρονται, η διακοινοβουλευτική συνάντηση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και Νοτιού Αφρική θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Ίσως να σας ε, ενδιαφέρει να παρευρεθείτε. Θα γίνει μια ενημέρωση για το που βρισκόμαστε στο COP17. Και όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στην διακοινοβουλευτική συνάντηση, και για αυτό το θέμα, αλλά και για τα άλλα συναφή ζητήματα, φυσικά να έρθουν. Και θα χαρώ να σας ενημερώσω μέσω του γραφείου μου ή μέσω της γραμματείας. Θα συζητηθεί και το θέμα του COP17. Φυσικά οι προσδοκίε μας είναι υψηλέ. Είναι ότι ο Αφρικανή φαίνεται να είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι. Αλλά πάντα τα δύο μεγάλα ερωτηματικά είναι η συμβολή και συμμετοχή των ήπα και της Κίνας. Αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να βγούμε με μια συμφωνία από την COP17. Και αν δεν είναι διεθνής αυτή η συμφωνία, δεν πειράζει. Αρκεί να υπάρχει ηγεσία στο θέμα αυτό και αυτό δεν χωράει άλλη καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιο άλλο να μιλήσει. Η Κομισιόν μήπω θέλει να πάρει το λόγο. Euh, Σα υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 4η Οκτωβρίου στι 12 το μεσημέρι και ότι πρέπει να υποβληθούν μόνο στα αγγλικά. Γιατί μόνο στα αγγλικά. Γιατί έχουμε αυτή τη διακριτική μεταχείριση. Α, για ε, να προλάβουμε ουσιαστικά για χρονικούς λόγους. Ε, τώρα θα μιλήσουμε για την ανταλλαγή απόψεων για την ε, σχέδιο γνωμοδότησης ε, ε, περί της χρηματοδότησης προς το Αφγανιστάν. Κύριε Κάσμαν, δεν συμφωνείτε. την τελευταία αυτή ανακοίνωση που κάνατε, από ό,τι ξέρετε, η προστασία και ο σεβασμό των άλλων γλώσσων στο θεσμικό όργανο αυτό είναι κάτι το ουσιώδες. Δεδομένης λοιπόν της κατάστασης ότι χρειαζόμαστε τις τροπολογίε στα αγγλικά, θα ήθελα να θεωρώ ότι όσοι δεν έχουν άνεση στα αγγλικά θα λάβουν μια μετάφραση από την σχετική υπηρεσία. Ιδάλλως, μπορεί να βρεθούμε σε μια θέση όπου σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε άτομο θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη συνέχιση της διαδικασίας, καθότι δεν θα υπάρχει μετάφραση των τροπολογιών στη γλώσσα τους. Ε, ελπίζω, ελπίζω να μπορέσουν να έχουν την υπηρεσία αυτή της μετάφρασης. Συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Παρά τις προσπαθίες μου να μάθω αγγλικά δυσκολεύομαι ακόμη πάρα πολύ. Είναι, μου είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να μου λένε ότι χρειάζονται 10 ημέρες για τη μετάφραση και ότι ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Είτε λοιπόν κατεβαίνουμε σε διαδήλωση είτε υποκύπτουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι φυσιολογικό, αλλά πρόκειται για ένα ζήτημα που εμφανίζεται διαρκώς. Εμεί το δεχόμαστε πρόβατα και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Αν θέλετε λοιπόν να οργανώσετε μια επανάσταση, θα συμμετέχω και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη κύριε Πρέντα, ε, μαζί με όλη την ομάδα. Εγώ, η αλήθεια είναι, δυσκολεύομαι τρομακτικά μου. Είναι τρομακτικά δύσκολο. Αποφάσισα την επόμενη φορά λοιπόν θα έχουμε μια κατεπίγουσα ψηφοφορία στα αγγλικά. Δεν θα συμμετέχω γιατί... Τώρα θα μιλήσουμε για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ε, σχέδιο γνωμοδότηση για το δημοσιονομικό έλεγχο τη χρηματοδοτική συνδρομή τη ΕΕ στο Αφγανιστάν. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου θα ψηφίσει τον Νοέμβριο μια έκθεση που παρουσιάζει μια κριτική ανάλυση των διαφόρων τρόπων χρηματοδότηση που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν, όπως και η συνδρομή που παρέχεται μέσω των μέσω πολλών ταμείων. Μιλάμε για τον έλεγχο, για τον συντονισμό μεταξύ χρηματοδοτών στο πολύ ευαίσθητο περιβάλλον του Αφγανιστάν. Δίνω τον λόγο στον κύριο Γκέρενς που είναι ο εισηγητής θα μας προσθέσει το σχέδιο γνωμοδότησης που αφορά τη συνδρομή της Επιτροπής ΔΕΒΕ σε αυτή τη συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συμφωνώ με όσα μόλις είπατε. Έχω μπροστά μου την έκθεση του Δημοσιονομικού Ελέγχου όπου απαριθμούνται οι διάφοροι οδοί χρηματοδότησης που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν, υποστηρίζει τη διατήρηση μιας διαφοροποίησης των τρόπων χρηματοδότησης και των εταίρων όπου ο καθένας έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Πρέπει να υπενθυμίσουμε επίσης ότι η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου επιμένει στις περιορισμένες δυνατότητες των αυγανικών αρχών ελέγχου. Ο κίνδυνος διαφθοράς είναι αρκετά υψηλός όπως γνωρίζετε. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε κάθε τύπο διαφθορά στο Αφγανιστάν, απλά δεν πρέπει να πάμε ποτέ εκεί πέρα. Η Κομισιόν παρουσιάζει τη δύνατα σημεία των έργων, πολύ αργή αναφορά, πολύ ελλειπής πρόσβαση στα αποτελέσματα, ανησυχεί επίσης λόγω της περιορισμένη πρόσβαση στις εκθέσεις ελέγχου που δίνουν τα, οι οργανισμοί των ΗΕ στην, στην Κομισιόν. Θα ήθελα η Κομισιόν να η Επιτροπή να δώσει τη γνώμη της. Για ποιο λόγο υπάρχει τόση δυσκολία να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Γίνονται συστάσεις για τη βελτίωση της παρακολούθησης και του reporting των αναφορών ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και ο συντονισμός με τους υπόλοιπους δωρητές που βρίσκονται, χρηματοδότες που βρίσκονται εκεί. Περιμένω τον καφέ εδώ και μια μισή ώρα. Ο διπλανός μου θα έρθει σε εκεί. Καφέ παρακαλώ. Όπως φαίνεται σήμερα δεν μπορώ να εκφραστώ καθαρά. από τη μία πλευρά, αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, δεν πρέπει να πάμε καθόλου σε αυτή τη χώρα. Αν πάμε όμως, ε, γινόμαστε αντικείμενο κριτικής. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε λίγο πιο λεπτομερώς τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ε, τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σχέδιο δράσης για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Από το 2009 πρόκειται για ένα πλαίσιο ωφέλιμο αλλά υπερβολικά γενικό. Για να υποστηρίξω λίγο και την Κομισιόν, θα ήθελα να πω ότι οι δράσεις της ε, ε, λαμβάνουν χώρα σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και επιτόπου. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου ζητά ε, να είμαστε προσεκτικοί να προσφύγουμε προσεκτικά στο τομεακό δημοσιονομικό, στη τομεακή δημοσιονομική υποστήριξη στο Αφγανιστάν. Ξέσπασε ένα σκάνδαλο. Βλέπουμε μια... Ε, Σταλθήκαν πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια από την Καμπούλ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και επίσης ανακαλύψαμε ότι ο, εμπλεκόταν ο αδελφός του Προέδρου. Η τράπεζα της Καμπούλ ε, δεν έκλεψε κανείς χρήματα που προήλθαν από την Κομισιόν, αλλά η τράπεζα της Καμπούλ ε, δεν είναι μια τράπεζα που δεν έχει κανένα σχέση με το κράτος. Από αυτή την άποψη το Αφγανιστάν με τα σκάνδαλά του επιδεινώνει την κατάστασή του. Όλοι έχουν ειδοποιηθεί, έμαθαν για αυτό το σκάνδαλο, το οποίο δεν αποτελεί το αντικείμενο της εκθεσής μου, αλλά πρέπει να το επισημάνω για να περιγράψω λίγο τις συνθήκες ε, υπό τις οποίες συντάσσεται αυτή η έκθεση. Γνωρίζουμε επίσης ε, ότι η στρατιωτική πτυχή θα έχει όλο και λιγότερη σημασία. Ε, διάφορες χώρες θα αποσυρθούν σιγά σιγά. Ήδη έχουν δοθεί προθεσμίες για την αποσύρσή τους. Γνωρίζουμε επίσης ότι το Αφγανιστάν δεν μπορεί να πετάξει με δικά του φτερά ακόμη. Αυτό, για να το πούμε καθαρά, σημαίνει ότι θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να έχουμε παρουσία. Μπορούμε, πιστεύω, να δεχθούμε τη σύσταση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, να ε, προσφύγουμε σε τομεακή ε, δημοσιονομική διαδικασία δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Εάν το ελεγκτικό συνέδριο κρίνει ότι είναι πολύ λίγα τα έργα τα οποία γίνονται υπό τον έλεγχο της Κομισιόν, μπορούμε φυσικά να ενημερωθούμε για αυτή την κριτική, αλλά είναι να την πάρουμε σοβαρά Πρέπει να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί στην Κομισιόν το απαραίτητο προσωπικό ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει αυτές τις εργασίες. Γνωρίζουμε το σκάνδαλο που ε, είχε λάβει χώρα την Κομισιόν στη δεκαετία του 90. Δεν της είχαν δοθεί όλα τα μέσα σε ανθρώπινους πόρους που χρειαζόταν η Κομισιόν ώστε να επιτύχει αυτά τα έργα. Είτε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτύξει ε, από μόνη της ε, τα έργα και θα πρέπει να της δώσουμε το σωστό προσωπικό ή θα πρέπει να απέχουμε οποιαδήποτε κριτική. Το Αφγανιστάν λοιπόν ε, έχει να αντιμετωπίσει μια γιγάντια πρόκληση. Δεν θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι Έχουν πετρελαϊκούς και ορυκτούς πόρους εξαιρετικά σημαντικούς Συνεπώς ε, όλος αυτός ο πλούτος ε, θα επανέλθει στα χέρια των αρχών αυτής της χώρας. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να συνοδεύουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που συνεχίζει να αποτελεί τον σημαντικότερο εγγυητή, χρηματοδότη, έχει μια πολύ ιδιαίτερη ευθύνη αν θέλουμε αυτή η χώρα να έχει κάποια ευκαιρία ε, για το μέλλον θα πρέπει να διατηρήσουμε τη βοήθεια και να προσαρμόσουμε τα έργα και τα προγράμματα στις ε, συνθήκες ε, να προχωρήσουμε περισσότερο στην τομεακή ανάπτυξη εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες να στηρίξουμε επίσης τους μη κυβερνητικού οργανισμούς. Πιστεύω ότι μόνο το έργο αυτών των μικρών στο Αφγανιστάν από μόνο του το έργο αυτό ε, αποτελεί το αντικείμενο συζήτησης επειδή εάν οι κυβερνητικές αρχές αποσυρθούν κάποιος θα πρέπει να πάρει τη σκητάλη. Αυτές είναι ουσιαστικά παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω. Όπως είπα στις εισαγωγικέ παρατηρήσεις μου δεν πρόκειται για το πιο εύκολο φάκελο και θα πρέπει να δράσουμε πολιτικά όπως σας περιέγραψα στην παρουσίασή μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέρενς. Κύριε Μπέργκμαν, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με ό,τι είπε ο Σαρλ Γκέρενς και νομίζω ότι η έκθεσή του θα συμβάλλει σημαντικά και στην έκθεση του συναδέλφου από την Επιτροπή Έλεγχου του Προπολογισμού. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια σημεία πολιτικής ε, φύσεως. Από το 2001 μόνο οι ΙΠΑ έχουν χαλάσει 57 δις δολάρια στο Αφγανιστάν. 57 δισεκατομμύρια δολάρια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δεν ξέρω τα ακριβή αριθμητικά στοιχεία, αλλά νομίζω ότι είναι γύρω στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέσα σε μια δεκαετία. Όχι, 75 λοιπόν στην Αυστραλία. 100 ας πούμε δις Πρόκειται για ένα απίστευτο χρηματικό ποσό προς μία χώρα μόνο. Και η βοήθεια αυτή, αν δει κανεί και τα αποτελέσματα, αν δει την προπαγάνδα που λέει υπάρχουν πολύ περισσότερα κορίτσια στα δημοτικά σχολεία σήμερα, ότι υπάρχει πρόοδο στον τομέα της υγείας. Ίσως να είναι και αλήθεια, αλλά για 100 δισεκατομμύρια δολάρια νομίζω θα μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω. Θα μπορούσαμε ίσω να έχουμε δώσει μια επιταγή σε κάθε Αφγανό. Θα ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να εμποδίζει τα χρήματα να φτάσουν εκεί που πρέπει. Έχουμε τρομερή ανασφάλεια, κάτι το οποίο επιδεινώνεται παρά την προπαγάνδα. Ε, είδαμε χθες ε, την επίθεση στο επίκεντρο της Καμπούλ, ε, στο πιο ασφαλή συνοικία. Δεν υπάρχει πιο προστατευμένη συνοικία κατά του πρώην Πρόεδρου Ραμπάνη. Πέραν της ανασφάλειας υπάρχει διαφθορά διαφθορά που επιδεινώνεται και αυτή η διαφθορά δεν υπήρχε πριν φτάσει η διεθνή κοινότητα. Η διεθνή κοινότητα έφτασε στο Αφγανιστάν το 2001 γιατί οι Ταλιμπάν είχαν πολλά ελαττώματα αλλά ο απολυταρχικός έλεγχος που είχαν στην συμπεριφορά και τη ζωή των πολιτών είχε ως πλεονέκτημα την πολύ περιορισμένη διαφθορά. Από το 2001 όμως και μετά έχει γίνει αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα η διαφθορά γιατί έπρεπε πάση θυσία να βρεθούν εταίροι, συνεργάτες ε, στον αγώνα κατά τον Ταλιμπάν. Ο Καρζάη ε, από διεφθαρμένους πρώην πολέμαρχους και ε, λαθρεμπόρους ναρκωτικών, ε, άτομα πραγματικά ανήθικα και τελικά δέχθηκε ε, η διεθνής κοινότητα να υπάρχει αυτή η ανομία στην κεφαλή του Αφγανιστάν. Και έτσι είχαμε στρεβλά αποτελέσματα, είχαμε τιμές παράλογες για το οτιδήποτε, είχαμε μισθούς πολύ υψηλότερους για αυτούς που εργάζονται για τη διεθνή κοινότητα, σε σχέση μας που δεν εργάζονται για τη διεθνή κοινότητα, για Αμερικάνους, Ευρωπαίους και λοιπούς, κάτι το οποίο έχει καταστροφικά αποτελέσματα και συνέπειες για την αφγανική κοινωνία. Και σε αυτό το πλαίσιο, το δηλητηριασμένο αν θέλετε, το μολυσμένο, έχουμε τώρα να συζητήσουμε τον έλεγχο των δαπανών. Πολύ ωραία λόγια είναι αυτά και σημαντικό είναι να πούμε ότι ε, η βοήθεια η δημοσιονομική, η τομεακή ή όχι τομεακή ε, μπορεί να παρασχεθεί με βάση πολύ αυστηρά κριτήρια σε ό,τι αφορά τους στόχους ε, και σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις και τους υπολογισμούς που κάνουμε για να διαπιστώσουμε αν είναι αποτελεσματικά ή όχι τα κονδύλια, όλα αυτά είναι ωραία και σημαντικά. Αλλά θα έχουν αποτέλεσμα μόνο εφόσον είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε να στηρίξουμε την ανεξαρτησία του αφγανικού δικαστικού συστήματος. Πρώτο αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει σε αυτό, είναι προτεραιότητα και πολύ σωστά. Και το δεύτερο είναι η ανεξαρτησία του ελεγκτικού συνεδρίου του Αφγανιστάν. Είναι με ένα αποτελεσματικό όργανο, αλλά δεν έχει εξουσίες πολλές. Και ο ίδιος ο Αφγανός πρόεδρος ε, είναι αυτός ο οποίος ε, θέτει τέρμα σε κάποιες έρευνες ε, όταν αυτές αφορούν φίλους του πρόεδρου Καζάη. Πρέπει να το πούμε αυτό. Το ξέρουν άπαντες. Ουδής όμως δραστηριοποιείται. Επομένως, πρέπει να γίνει αυτή η πολιτική επιλογή, δηλαδή να ε, καταπολεμηθεί η διαφθορά στο κέντρο του κράτους. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, πρώτα απ' όλα ποτέ δεν θα είναι αποτελεσματική η βοήθεια, αλλά ποτέ επίσης δεν θα υπάρχει και η νομιμότητα, η νομιμοποίηση των αρχών στο Αφγανιστά στα μάτια των πολιτών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλει το Αφγανιστάν κάποια στιγμή να επιβιώσει και να προχωρήσει μόνο του χωρίς εμάς. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί στην έκθεση και γι' αυτό θα υποβάλω και σχετική τροπολογία σήμερα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέρμαν για τα πολύ σοφά σας λόγια. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον εισηγητή. Υπό το βλέμμα των όσων είπαν οι συναδελφοί μου, το ζήτημα είναι ότι συζητάμε για αυτή τη συνδρομή προς το Αφγανιστάν αμέσως μετά την ψηφοφορία της έκθεσης που εγώ συνέταξα για την αποτελεσματικότητα της ε, βοήθειας. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ε, πτυχή αυτή της αποτελεσματικότητας της βοήθειας για την οποία μόλις ψηφίσαμε σε αυτή την πολύ συγκεκριμένη περίπτωση όπως ήδη ακούσαμε εδώ πρόκειται για μια σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υπάρχουν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι που μόλις περιέγραψαν οι συναδελφοί μου. Εγώ θα προσέθετα μερικά σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε με τροπολογίες ε, ε, σε σχέση στην ε, γνωμοδότηση που έχει υποβλήθει. Πιστεύω ότι πρέπει να επισημανθεί το γεγονό ότι η βελτίωση των δυνατοτήτων της αφγανικής κυβέρνησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και κυρίως ε, των δομών που μπορούν να, να εξασκήσουν ε, λειτουργία επίβλεψης ε, θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Όπως είπαν οι συναδελφοί μου, θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών που θα μπορούσε να προειδοποιεί για περιπτώσεις διαφθοράς. Επίσης θα ήθελα να επισημάνουμε τη συνεργασία με τους υπόλοιπους δωρετές η οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί. Και πάλι στο τομέα, στον έλεγχο των μηχανισμών που θα μπορούσαν αν μη τι άλλο να βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε ένα κομμάτι της διαφθοράς Επίση, ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση στην Κομισιόν, αν είναι δυνατόν. Τέλος Δεκεμβρίου του 2010 υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα για το Αφγανιστάν και σε αυτό το ψήφισμα αναφέρονταν ε, λύσεις ε, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ε, ευθύνης σε ζητήματα χρηματοοικονομικής βοήθειας. Αναφέρω κυρίως ε, την ιδέα δημιουργίας μιας αποκεντρωμένης βάσης δεδομένων σε σχέση με ε, το αντίκτυπο της βοήθειας και επίσης ε, προτάθηκε να γίνει μια ευρεία μελέτη για το αντίκτυπο των χρηματοοικονομικών έργων. Ήθελα να μάθω αν έχουμε σημειώσει προόδους σε αυτά τα στοιχεία του ψηφίσματος που ψηφίσαμε στα μέσα Δεκεμβρίου του 2010. Μπορεί λοιπόν η Επιτροπή να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τους το ρωτήσουμε σε λίγο. Δίνω το λόγο στον κύριο Κάσμαν πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστώ. Φυσικά απόλυτα υποστηρίζω την προσέγγιση του κυρίου Γκιουρέντς. Ακούω και τι λένε οι συνάδελφοι αλλά να κάνω κάποιες μικρές σημειώσεις στα θέματα διαφάνειας και υπολογοδοσίας θα πρέπει να ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Να μην εξαιρέσουμε, αν θέλετε, και ξεχωριστά να φέρουμε το Αφγανιστάν, γιατί άλλως θα αποσταθεροποιηθεί αυτή η σταθερότητα την οποία επιδιώκουμε. Επίσης, να θυμόμαστε ότι τα προβλήματα του Αφγανιστάν προέρχονται ε, αν θέλετε, και από μια περίοδο πριν από 250 χρόνια, μεταξύ άλλων και για, λόγω της Βρετανικής ε, ανάμειξης των 19ο αιώνα. Και κοιτώντας την ιστορία της χώρας, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε το Αφγανιστάν, που θεωρώ ότι βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκαιρία. Η ίδρυση και η υποστήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων για την καλύτερη κυβέρνηση αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο και πιστεύω ότι πλέον είναι καιρός να μην αμφισβητούμε τη δεσμευσή μας στο Αφγανιστάν. Όχι, να την επαναεπιβεβαιώσουμε, να την υπογραμμίσουμε, γιατί βλέπουμε αλλαγές και εξελίξεις και μετά γίνονται πάρα πολλά βήματα προς τα πίσω. Ε, οι μάχες μεταξύ των φυλών στην Καμπούλ και στην υπόλοιπη περιοχή. Όλα αυτά σημαίνουν ότι θα πρέπει να συνεχίσει την δέσμευση της η Ευρωπαϊκή Ένωση μια εποχή που οι άλλοι, αν θέλετε, διστάζουν και περιμένουν και την υπαναχώρηση της ε, παροχής δωρεών προς το Αφγανιστάν. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι θα γίνει και μακροπρόθεσμα. Ναι, διανύουμε μια εποχή οικονομικών προβλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, αλλά αυτό δεν συγκρίνεται καν με το τι συμβαίνει στο Αφγανιστάν και σε άλλες χώρες και το τι έχουν περάσει αυτές οι χώρες εδώ και αιώνες, κυρίως λόγω της απεικιοκρατίας. Ευχαριστούμε κύριε Κάσμαν. Η κυρία Θεοχάρους έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ολόκληρη η διεθνής κοινότητα και κυρίως αυτοί που είχαν άμεση εμπλοκή στο ζήτημα του Αφγανιστάν κοίταζαν μόνο το Αφγανιστάν και ποτέ τους Αφγανούς. Γι' αυτό έχει παρατηρηθεί και αυτή η τρομακτική αποτυχία των διεθνών σχέσεων όσον αφορά την περίπτωση αυτή, που είναι ιδιάζουσα περίπτωση και γι' αυτό θα έλεγα ότι ναι, η έκθεση του κυρίου Πρέτα μπορεί να είναι πολύ σημαντική για την τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της διεθνούς βοήθειας, αλλά για την περίπτωση του Αφγανιστάν θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε ξεχωριστά κριτήρια. Στηρίζω την έκθεση του κυρίου Γκέρενς, ε, είναι πάρα πολύ σημαντική, ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε και ίσως να το κάνουμε με τροπολογίες ότι δεν έχουμε καταφέρει καθόλου να αντιμετωπίσουμε την διαφθορά σε κανένα επίπεδο. Η ηρωίνη η οποία παράγεται στο Αφγανιστάν μαζί με την ηρωίνη στην κοιλάδα του ποταμού Τσου στο Τσου Βαλί εξακολουθεί να είναι η καλύτερη ποιότητα και σε τεράστιε ποσότητε ίσω το 90% τη παγκόσμια παραγωγή που έρχεται προ την Ευρώπη. Η κατάσταση των γυναικών δεν έχει βελτιωθεί καθόλου από το 1995 που αν θυμάστε κάποιοι είχε υπάρξει μια τρομακτική εξέγερση σε όλη την Ευρώπη Raise the veil from the Afghan women. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή την ιστορία. Ούτε η κατάσταση των παιδιών έχει βελτιωθεί και πολύ περισσότερο η κατάσταση των ηλικιωμένων. Οι σχέσει των ανθρώπων εξακολουθούν να είναι στο επίπεδο που ήταν προηγουμένω, δηλαδή αν σε μια οικογένεια δεν υπάρχει κάποιο άντρα για να φέρει την ανθρωπιστική βοήθεια στο σπίτι, η οικογένεια εξακολουθεί να πεθαίνει από την πείνα και οι γυναίκε ελάχιστε δυνατότητε έχουν να πηγαίνουν στο σχολείο. Τώρα, όσον αφορά τι NGOs, τι μη κυβερνητικέ, εμένα να μου επιτρέψετε να πιστεύω ότι οι πιο πολλέ από αυτέ είναι οίκιστα κυβερνητικές, δηλαδή ε, ε, είναι στην πραγματικότητα το μακρύ χέρι του κράτους και με αυτόν τον τρόπο γίνεται σημαντικός έλεγχος της βοήθειας. Μην ξεχνάτε και πόσοι ξένοι έχουν δολοφονηθεί γιατί είχαν κάποιες σχέσεις με περίεργες μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Γι' αυτό το λόγο θα έλεγα ότι εφόσον τόσα πολλά δισεκατομμύρια διοχετεύονται σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να, να κατανοήσουμε ότι ο τρόπος που διοχετεύονται σίγουρα δεν είναι αποτελεσματικός και να ψάξουμε ένα καλύτερο τρόπο για να ελέγχουμε παραγνωρίζοντας τις περιστασιακές κυβερνητικές σχέσεις και τις κυβερνήσεις του Αφγανιστάν που είναι βουτυγμένες μέσα στη διαφθορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριος ναι, θα ήθελα να προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε. Φυσικά και στηρίζω απόλυτα αυτό που είπε ο Μάικλ Κάσμαν. Η δέσμευσή μα στο Αφγανιστάν ε, δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί επειδή προβαίνουμε σε αυτές τις τρομερές διαπιστώσεις. Ε, το αντίθετο, απλά θα πρέπει να βγούμε από αυτές ε, τις καταστροφικές χρονιές της εποχής Μπούς. Έχω ένα ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, προς την Κομισιόν. Μας έχουν προειδοποιήσει ότι επίκειται λοιμός ε, στο Αφγανιστάν λόγω της ε, ξηρασίας ε, που θα απειλήσει μάλλον σύμφωνα με την Oxfam 3 εκατομμύρια άτομα. Αυτή είναι η έκθεση της Oxfam αυτής της εβδομάδας. Το έχει υπόψη της Κομισιόν και τι προτίθεται να πράξει γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Είναι πάντως μια ακόμη απόδειξη της αναποτελεσματικότητας της βοήθειας που δαπανάται. Merci beaucoup. Je passe... Ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στην Κομισιόν. Κυρία Τζινάρο η κυρία Κολέκα ή κυρία Κώστα. Όπως θέλετε. Ε, good morning. Thank you very much for... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους βουλευτές για τα πολύ χρήσιμα σχόλια, τα οποία εκτιμούμε ιδιαίτερως. Εκτιμούμε την ανεξάρτητη οπτική γωνία που συμβάλλει στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και, το, και η οποία βελτιώνει τον τρόπο εργασίας μας και μας βοηθάει να βοηθήσουμε να βελτιώσουμε την εργασία μας και με τους άλλους δωρητές. Να υπογραμμίσω τώρα κάποια στοιχεία και αν θέλετε φυσικά να επισέλθω και σε λεπτομέρειες για να εξηγήσω καλύτερα. Αυτό μπορεί να γίνει και εκ των υστέρων εγγράφος, αν προτιμάτε. Να σημειώσω ότι το Αφγανιστάν, όπως αναφέρεται ήδη, είναι σε μια μεταβατική φάση μεταξύ τα χρόνια των, των χρόνων σύγκρουσης, μετά τα χρόνια σύγκρουσης και μετά τις εσωτερικές συγκρούσεις, με όλες τις θεσμικές αδυναμίες που συνδέονται με αυτό και σε ό,τι αφορά τους κινδύνους για την εφαρμογή της αναπτυξιακής βοήθειας. Θα πρέπει αυτή την πραγματικότητα να την αναγνωρίσουμε. Σε αυτή την κατάσταση παρέχει την βοήθεια της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι άλλοι δωρητές. Επίσης, να υπογραμμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί μια προσέγγιση μακροπρόθεσμης δέσμευσης και προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε αφενός την ανάγκη να υπάρχει μια χώρα όπου θα πληρούνται οι άμεσες ανάγκες του πληθυσμού σε ό,τι αφορά την υγεία, για παράδειγμα, και τις κοινωνικές ε, υπηρεσίες, αλλά παράλληλα αφετέρου θα υπάρχει και ε, μία παρακολούθηση της γενικότερης βελτίωσης και μακροπρόθεσμης βελτίωσης της διακυβέρνησης σε περιφερειακό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο και της θεσμικής βελτίωσης ε, Στου τομεί τομείς οποίου οποίους δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δικαιοσύνη και το καθεξή. Όντως, πολλά κονδύλια έχουν δαπανηθεί στο Αφγανιστάν από τους διεθνείς διοριτέ μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δαπανίσει 1,8 δις θα πρέπει ασφαλώς να υποστηρίζουμε τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και τις πολιτικές της κυβέρνησης μεταξύ των οποίων και η θεσμική ανάπτυξη. Εστιαζόμαστε σε κάποιους τομείς όπου βλέπουμε ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλουμε πάντα να υπάρχει η κατανομή των εργασιών μεταξύ των δωρητών. Όντως, ο κατακαιρματισμός ε, των δωρεών στο Αφγανιστάν και η αποτελεσματικότητα της ε, αρρωγής δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Και αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Καταρχάς, ε, πολλοί δωρητές, πολλές χώρες που εμπλέκονται και στρατιωτικά έχουν στρατιωτική παρουσία. Σημειώνεται κάποια πρόοδος, ωστόσο πολύ αργή. Το παραδέχομαι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πρόοδος είναι σημαντική. Η πρόοδος των τελευταίων δύο ετών. Σε ό,τι αφορά το συντονισμό της βοήθειας μετά την έγκριση του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αφγανιστάν γίνονται εξαμηνίες εκθέσεις τακτικά οι οποίες και συζητιώνται στο Συμβούλιο και εγκρίνονται από το Συμβούλιο μάλιστα. Συμφωνούμε απόλυτα ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η εθνική κυβέρνηση, οι θεσμικοί οργανισμοί και οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνε για την οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό είναι πέρα από κάθε ε, αμφιβολία. Επίσης, σε μεγάλο βαθμό ε, αντικαθιστάται, υποκαθιστάται ε, η λειτουργία των ε, εθνικών υπηρεσιών από τους διεθνείς δωρητές μέσω της τεχνικής βοήθειας το οποίο επιτρέπει να συνεχίζουν κάποιες πολιτικές, αλλά τίθεται το ερώτημα του κατά πόσο είναι βιώσιμη αυτή η προσέγγιση μακροπρόθεσμα. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μετάβαση και την περίοδο μετά το 2014. τα δύο βασικά ζητήματα που θα συζητηθούν στην Βόνη το Δεκέμβριο. Να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στις προπαρασκευαστικές εργασίες της ε, Συνόδου της Βόνης. Τώρα, η επιλογή των στοιχείων εφαρμογής. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει να κάνει και με το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε. Γι' αυτό το λόγο και μόνο χρησιμοποιήσαμε την κεντρική, όπως λέμε, διαχείριση. των συμβάσεων. Δεν επιτρέπουμε δηλαδή στους Αφγανούς να διαχειρίζονται τις συμβάσεις λόγω των κινδύνων που ενέχονται. Αυτό το κάνουμε στον τομέα της υγείας. Ωστόσο, οι έλεγχοι μας ε, κατέδειξαν ότι δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα θέλαμε. Ελπίζουμε ότι το νέο πρόγραμμα για την υγεία θα μας επιτρέψει τουλάχιστον να κινηθούμε προς μία ε, προσέγγιση που θα καλύπτει όλους τους τομείς. Τώρα, ένας άλλος τομέας που επιλέξαμε για την τεχνική μας αρρωγή είναι η χρήση των ε, ταμείων από πολλαπλούς δωρητές, όπου ενώνουμε, αν θέλετε, τις δυνάμεις μας με τους Ιάπωνες και άλλους δωρητές. Έχουμε κάνει και πολλές προσπάθειες για να ενισχύσουμε και την ανιστομία και θα πρέπει να πούμε ότι χάρη στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταφέραμε να τα μεταρρυθμίσουμε τα trust funds αυτά. όχι μόνο για την μισθοδοσία των αστυνομικών, αλλά και για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής διακυβέρνησης στον τομέα αυτό. και θα θέλαμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της υποστήριξης του υπολογισμού του προπολογισμού. Χρειάζονται φυσικά οι απαραίτητοι όροι σε ό,τι αφορά την ικανοποιητική δημοσιονομική διακυβέρνηση. Δεν χρειάζεται να είναι τέλεια, αλλά θα πρέπει να μας εμπνέει εμπιστοσύνη. για αποφυγή και πρόληψη καταχρήσεων και άλλων απατών. Θα πρέπει να υπάρχουν επίσης και άλλες στρατηγικές και άλλοι όροι οι οποίοι θα πρέπει να πληρούνται. Προτού κινηθούμε προς την άμεση υποστήριξη του υπολογισμού. Θα σταματήσω στο σημείο αυτό. Αν θέλετε, Ασφαλώς θα σας δώσουμε και επιπλέον πληροφορίες, είτε εδώ στην συνάντηση, είτε και αργότερα γραπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Γκέρεντς για να ολοκληρώσουμε. Συγγνώμη, δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε. Θέλετε να ξανακάνετε την ερώτησή σας. Με συγχωρείτε κύριε Γκέρεντς. Συγγνώμη, θα ήθελα απλά να επιμείνω. Δεν μας λέτε τίποτα για το πρόβλημα της ξηρασίας που, ε, για το οποίο έκανα μια ερώτηση. Ε, Η Κομισιόν θέλει να απαντήσει όσον αφορά το ζήτημα της ξηρασίας είναι πρόσφατες πληροφορίες η άμεση απόκριση στη ξηρασία αποτελεί ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα είμαστε λοιπόν σε επαφή με την DG ECO και θα δούμε πως η Κομισιόν θα μπορούσε να αποκριθεί στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης υποστήριξης θα επαναλάβω ότι ένας από τους τομείς εστίασης ε, για τη συμμετοχή και την αρρωγή της Κομισιόν στο Αφγανιστάν είναι η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη. Αυτός ε, ο τομέας ε, καταλαμβάνει μεγάλο κομμάτι της αρρωγής μας. Υποστηρίζουμε τη βελτίωση των συστημάτων άρδευσης που ελπίζουμε στο μέλλον θα βοηθήσει στην ε, πρόληψη ή τουλάχιστον στο μετριασμό των επιπτώσεων ε, ενδεχόμενης ξηρασίας, ε, θα βελτιώσει τις τεχνολογίες παραγωγής στον τομέα της γεωργίας, εκπαίδευση επίσης και επίσης οι υπηρεσίες που παρέχονται στους αγρότες. Σχετίζεται επίσης με το ευρύτερο πρόγραμμα υποστηρίξης της αγροτικής ανάπτυξης. Ε, συνεργαζόμαστε με ΜΚΟ και τώρα ε, προσπαθούμε να βρούμε συγκεκριμένε οδούς μέσω εθνικών προγραμμάτων, μέσω του ΑΕΡΤΙΕΦ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Γκέρενς για, το, για να μας πει τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, που μίλησαν για την εκθεσή μου. Ευχαριστώ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες τους. Αναμένω τις τροπολογίες που θα υποβάλουν. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που ήθελα να πω, ε, πιστεύω ότι αυτό βλέπουμε κοινό σε όλες τις ομιλίες που ακούσαμε. Η διακυβέρνηση στο Αφγανιστάν αποτελεί ευθύνη του Αφγανιστάν. Θα πρέπει λοιπόν να μείνουμε στο πλευρά τους. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο χρόνος πιέζει ε, όπως ξέρουμε θα αλλάξει η κατανομή της αρρωγής του Αφγανιστάν στο μέλλον. Οι ομάδες ανοικοδόμησης επαρχιών έχουν διασφαλίσει περιοχές όπου μπορούμε να παρέχουμε αρρωγή. Εκεί θα πρέπει να αναπτύξουμε και να επινοήσουμε ένα άλλο είδος ε, συνδρομής, ένα άλλο είδος συνεργασίας. Είχα προτείνει μεγαλύτερη συμμετοχή τον ΜΚΟΕ μικρόν αυτό όμως θα πρέπει να γίνει με ασφάλεια. Θα πρέπει να συμβάλλουμε λοιπόν στην ανάπτυξη των δυνάμεων τάξης στο Αφγανιστάν. Σε 10 Αφγανούς, 2 ε, ή 3, ε, σε 10 Αφγανούς 2 ή 3 μπορεί να συμμετέχουν, ε, να συνεργάζονται με τους Ταλιμπάν. Κανείς δεν έχει μπορέσει μέχρι σήμερα να μου εξηγήσει τι είναι ένας Ταλιμπάν ε, θα ήθελα επίσης ε, να δούμε και τα θετικά σημεία. Υπάρχουν γυναίκες στο Αφγανιστάν που σηκώνουν το κεφάλι. Πόσο αξίζει μια γυναίκα που έχει το θάρρος να επιβληθεί, να αναπτυχθεί, να μορφωθεί, να πάνε... τα κορίτσια που πάνε στο σχολείο είναι κάτι που δεν υπήρχε πριν. Αυτό πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι ένα από τα πράγματα που εμείς προσφέραμε. Η διεθνής κοινότητα προσέφερε. Η Καμπούλη επίσης πολύ έχει αλλάξει εκ Δεν, ε, είναι μια πόλη πια που δεν έχει ζωή μόνο σε ένα δρόμο, έχει αλλάξει ριζικά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ε, αυτός είναι και ένας οικονομικός παράγοντας τρομακτικά σημαντικός σε μια χώρα όπου ελέγχεται ίσως όχι όλοι αλλά από κεντρική κυβέρνηση δεν ξέρουμε αν θα κερδίσουμε τα στοιχήματα. Ξέρουμε ότι θα χάσουμε. Όμω, εκ των προτέρων, αν φοβόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε σε θέματα διακυβέρνηση όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Θα πρέπει να είμαστε έξυπνοι και να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας ώστε να αναπτύξουμε έξυπνες συνεργασίες και εταιρικέ σχέσεις με το Αφγανιστάν. Αυτή η άποψη της Κομισιόν είναι άψογη, έχουν κάνει εξαιρετικό έργο Πρέπει επίσης να δείξουμε σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή τη χώρα, να μην σε αυτή τη χώρα όπου κανείς δεν ταξιδεύει ως ε, τουρίστη, τουρίστας που αγόρασε βάουτσες στο κλαμπ με την Θα πρέπει επίσης ε, να λάβουμε υπόψη και τους υπόλοιπους εταίρους σε θέματα ανάπτυξης και ανθρωπιστικής ε, βοήθειας και οι οποίοι έχουν φέρει αποτελέσματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένας οργανισμός ε, στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών ο οποίος είναι υποδειγματικός και ο οποίος μπορεί να προσφέρει λύση στο Αφγανιστάν. Πρόκειται για το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τους πληθυσμούς. Ξεκίνησε στη... Διευθυνόταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ε, στο Αφγανιστάν από μια γυναίκα από τη Σαουδική Αραβία, εξαιρετική, η οποία από τη μια μέρα στην άλλη ε, βρέθηκε χωρίς καμία συμβολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή υπό την κυβέρνηση Μπούς την κατηγορούσαν ότι διαδίδει τις αμβλώσεις στην Κίνα, το οποίο δεν είναι αλήθεια. Ε, έγινε μια επιτροπή ερευνητική στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε πάρει ε, χρήματα τα οποία χρειαζόταν οπωσδήποτε για να προσφέρει κάποια βοήθεια στις γυναίκες του Αφγανιστάν προβλήματα τέτοιου είδους ε, πρέπει να τα μαθαίνουμε. Εγώ όταν ήμουν υπεύθυνο σε εθνικό επίπεδο είχαμε καταφέρει η Κομισιό να αποδεχθεί μια επιπλέον χρηματοδότηση για την απόσυρση των ΗΠΑ. Αυτός ο οργανισμός έκανε εξαιρετικό έργο. Επανέρχομαι στους ΜΚΟ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εμπλακεί σήμερα η Κομισιόν σε διαπραγματεύσεις που ε, δεν θα λάβουν χώρα με τους ε, τα Ταλιμπάν. Πιστεύω ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε επαρκές περιθώριο ώστε να διασφαλίσουμε τη δράση των ΜΚΟ. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις θα χρειαστεί να αναδείξουμε την αμεροληψία των ανθρωπιστικών οργανώσεων επειδή βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν τους Αφγανούς ε, οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις, κάπο μικρών αυτές δεν τους είναι ευχάριστο όλο αυτό που κάνουν δεν, τους είναι, δεν το κάνουν από ευχαρίστηση προσπαθούν να βοηθήσουν να προσφέρουν συμβολή με μόνο σκοπό την ανάπτυξη του αφγανικού πληθυσμού είναι κρίμα που αυτή η έκθεση είναι μόνο γνωμοδότηση. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα να πούμε και τόσε μικρέ ευκαιρίε να το κάνουμε, τόσε λίγε ευκαιρίε να εκφραστούμε. Πιστεύω και ελπίζω ότι το μήνυμά μα ε, έχει ε, βρει ε, ακροατέ στην Κομισιόν, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει κάνει εξαιρετικό έργο στο Αφγανιστάν. Ευχαριστούμε πολύ. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για την γνωμοδότηση αυτή Λίγη στις 23 Σεπτεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι. Και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 11 Οκτωβρίου. Λοιπόν, επόμενο σημείο. Τον Απρίλιο η Κομισιόν δημοσίευσε την ανακοίνωσή τη για τον τρόπο ενίσχυση ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα χρηματοδότηση τη ανάπτυξη. Αυτή η ανακοίνωση αναφέρει και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τα κράτη-μέλη σε σχέση με του στόχου τη χιλιετία, αλλά και άλλα σημαντικά θέματα. Επί παραδείγματι, η αποτελεσματικότητα της βοήθειας, μηχανισμοί καινοτόμοι, μηχανισμοί χρηματοδότησης, χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, παγκόσμια διακυβέρνηση. Εμείς αποφασίσαμε ως Επιτροπή να θέσουμε στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν μια προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια, θα συνοδεύεται και από ψήφισμα. Σχέδιο των κειμένων έχετε λάβει, και όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο των παραπαρασκευαστικών εργασιών για την διάσκεψη του Μπούζαν για την επιτελεσματικότητα της βοήθειας. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στην Κομισιόν για να μας παρουσιάσει την ανακοίνωσή της και εν συνεχεία στους βουλευτές θα το ήθελαν. Κυρία Άλεν είναι νομίζω η αρμόδια από την Επιτροπή, δεν ξέρω αν παρίσταται. Είναι εδώ κυρία Άλεν. Bonjour. Euh, Δυστυχώς δεν είχατε θέσει το ερώτημα στην ιστοσελίδα, άρα είμαι κάπως απροετοίμαστη να το πω. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα so the first question is, is it τεσσάρων τμήματων. Καταρχάς, ε, είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν οι δεσμεύσει της Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στους στόχους της. Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ κατά πόσο είναι ρεαλιστικό ή όχι. Αν οι ηγέτε τη Ευρωπαϊκής Ένωση έχουν ε, επιβεβαιώσει τη δέσμευση να πετύχουν του στόχους και το ίδιο έχει κάνει και το Συμβούλιο του Ιουνίου, τι να πω, φυσικά αποτελεί πρόκληση. Και έχουμε ήδη αναφέρει στους Υπουργούς ε, Ανάπτυξης τον Ιούνιο ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση ως έχει, φυσικά δεν πρόκειται να πετύχουμε τους στόχους. Δεύτερη ερώτηση. Από πού θα προέλθουν οι επιπλέον χρηματοδοτήσεις. Ε, τι βήματα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη για να βγάλουν αυτά τα επιπλέον κονδύλια. Τα χρήματα θα πρέπει να προέλθουν από τα κράτη-μέλη, από τους προπολογισμού τους. Άρα, ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να λάβει οποιαδήποτε βήματα πρότασης προς τα κράτη-μέλη για το πώς θα κινήσουν και θα κινητοποιήσουν τους πόρους της, αλλά αυτό που κάναμε είναι στις προτάσεις μας για τις επόμενες δημοσιονομικές πρακτικές είναι να, να προτείνουμε έναν φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτό θα αποτελέσει μια επιπλέον ε, πηγή πόρων που θα αφαιρέσει αν θέλετε κάπως, θα απαλύνει κάπως την πίεση που δέχονται τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τον άμεσο φόρο. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν και θα πρέπει να ξεκινήσουν οι συζητήσεις με το Συμβούλιο και με εσά. Μία τρίτη ερώτηση για μία εγγύηση για την κινητοποίηση καινούριων και παλαιών ε, φόρων και πόρων για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος προκειμένου να μην εκτραπούν αυτά τα κονδύλια Συμφωνώ απόλυτα με το αίτημα αυτό, αλλά φυσικά κάποια ζητήματα ανακύπτουν. Καταρχάς, η υποστήριξη προς, τα, προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για α, την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος μπορεί να θεωρηθεί ODA. Κατά δεύτερον, για τις επιπρόσθετους πόρους. Αυτό προέρχεται από τις, τις, ε, ε, τη Συμφωνία της Κοπενχάγης. Ωστόσο, δεν υπάρχει πουθενά ε, ορισμός για το τι σημαίνει καινούργιοι και επιπρόσθετοι πόροι και εκ παραλλήλου το Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει κατά πόσον οι πόροι γρήγορης κινητοποίησης αποτελούν επιπρόσθετους πόρους. Άρα, δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε κάτι πιο αυστηρό από αυτό που θα αποφασιστεί σε επίπεδο ε, oh Άρα και εδώ περιορισμένη συμβολή μας. Τελευταίο ερώτημα, το οποίο μάλλον δεν έχει να κάνει με την ίδια την έκθεση, έχει να κάνει με την συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην επόμενη περίοδο του ΩΣΑ σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια και την σχετική αναθεώρηση. Σας υπόσχομαι ότι θα συμμετάσχετε η διερευνητική αποστολή των ΔΑΚ, των ομοτήμων ΔΑΚ, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Η ημερομηνία διεξαγωγή τη επίσκεψη στι Βρυξέλλε θα είναι μισό λεπτό γιατί κάπου το έχω. Αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί μιλάει πάντα έτσι. 10 14 Οκτωβρίου και θα διοργανωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεχωριστή συνάντηση με τους ομοτήμους, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, για να τους γνωρίσετε. Και στην προηγούμενη άσκηση, το 2007, άλλωστε είχατε την ευκαιρία αυτή. Την ίδια λοιπόν πρόσβαση θα έχετε στην ομάδα των ομοτήμων, όπως και στο παρελθόν. Θα σταματήσω στο σημείο αυτό. Αν έχετε ερωτήσεις, ευχαρίστω να τις απαντήσω. Κοιτώντας το σχέδιο κειμένου, ωστόσο, βρήκα δύο λάθη, σφάλματα. να τα διορθώσουμε ίσως. Μία σύσταση στο πρώτο τμήμα, όπου γίνονται όλες οι αναφορές στα έγγραφα αναφοράς. Στην ομοφωνία γίνεται μία αναφορά, αλλά όχι στο επόμενο συνεδρίο της Ντόχα το 2008. Καλό νομίζω είναι να υπάρχει και αυτή η αναφορά Γιατί στην τρίτη παύλα από το τέλος αναφέρεστε στο ψήφισμά σας εν ώψη της διάσκεψης της Δόχα αλλά είχε λάβει ώρα η διάσκεψη της Δόχα. Αυτό λοιπόν αποτελεί μια μια πρώτη πρόταση αν θέλετε από μέρος μου και στο ένα καλώς ορίζετε την έκθεση, σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και ζητάτε από κάποια κράτη-μέλη να δημοσιεύσουν τις απαντήσεις τους. Όλα τα κρατη έχουν συμφωνήσει να δημοσιευτούν οι απαντήσεις τους. Το κάναμε αυτό, τα έχουμε βάλει και σε ε, ένα website, σε μια ιστοσελίδα και έχω στείλει και το σύνδεσμο στη γραμματεία. Άρα υπάρχουν αυτά online πλέον. Να σταματήσω στο σημείο αυτό, να πω ότι πολύ χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προετοιμάζει το ψήφισμα αυτό αυτό καταδεικνύει ότι είμαστε σύμμαχοι και ότι αγωνιζόμαστε για τον ίδιο στόχο. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν την Επιτροπή. Okay. Euh, simplement un petit Μια μικρή λεπτομέρεια. Θα ελέγξουμε όλα τα έγγραφα και τα σχόλια βρισκόνται στην τοποθεσία από την Τρίτη και διανεμήθηκαν και στο φάκελο που λάβατε στην είσοδο. Δεν υπήρχε σφάλμα από αυτή την άποψη. Χρειάζεται να κάνουμε μια συνεδρίαση με την Κομισιόν, με τον ΟΣΑ χωρίς την Κομισιόν. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή. Νομίζω ότι η επαφή θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα. Οι συνάδελφοί μου, οι αρμόδιοι, είχαν κάποιες επαφές ε, στη Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιου Τράπεζας που λαμβάνει χώρα αυτή τη εβδομάδα αλλά πιστεύω ότι θα επικοινωνήσει μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι αυτή είναι η σημαντικότερη συνάντηση που έχει την επόμενη εβδομάδα. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Κάσμαν Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Κομισιόν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Χρειαζόμαστε κάποια συμμαχία. Επειδή για πολύ καιρό αυτή η Επιτροπή επικροτεί τη δέσμευση για τη χρηματοδότηση, αλλά ανησυχεί επίσης ε, κατά πόσο τα κράτη-μέλη επιτυγχάνουν τη δεσμεύσή τους. Ε, αναφορές λοιπόν σε θέματα χρηματοδότησης είναι ζωτικά ώστε να υπάρχει ευθύνη των κρατών μελών. Σύμφωνα με την Κομισιόν χρειαζόμαστε να υπάρχουν πολύ σαφείς ορισμοί για οτιδήποτε νέο ή πρόσθετο. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι όσα μας υποσχέθηκαν στην Κοπενχάγη είναι κάτι πρόσθετο. Ε, σήμερα αυτό φαίνεται να το παραβλέπουμε. Χαίρομαι που αναφέρεστε στις διορθώσεις και επικροτούμε οποιασδήποτε διορθώσεις ε, αυτό σημαίνει ότι η προσέγγιση μας είναι ακριβής. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας για το ψήφισμά μας. Καλό είναι που αναφερθήκατε σε αυτό. Πιστεύω ότι έτσι αντιλαμβανόμαστε την ουσία του γιατί έχουμε υποβάλει προφορικές ερωτήσεις. Εάν δεσμευτούμε ή η Κομισιόν δεσμευτεί εκ μέρους μας και του Συμβουλίου όσον αφορά ένα στόχο, και μετά ξαφνικά μας λείπουν 50 δισεκατομμύρια από αυτό το στόχο, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε κάτι τέτοιο. Αν δεν μπορούμε να το διατηρήσουμε πρέπει συλλογικά να θέσουμε πίεση στα κράτη-μέλη ώστε να καλύπτουν τις δεσμεύσεις τους του 0,7 του ε, ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ε, Με εξαίρεση κάποιες χώρες, στο Βέλγιο, τη Σουηδία, καμία χώρα δεν φτάνει καν στο 0,6% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματο. Νομίζω ότι σε μέσο, κατά μέσο όρο τα κρατη το καλύπτουν κατά 0,3 ή 0,4. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις. Η 04 αυτο ειναι απαραδεκτο εχουμε να αντιμετωπισουμε κρίση η κριση της κλιματικής αλλαγής υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Και ξαφνικά μα ήρθε σαν να μην την γνωρίζαμε, σαν να μην την είχαμε ξαναδεί πριν από 6-7 χρόνια. Έχουμε δεσμεύσει του πόρου για να την αντιμετωπίσουμε. Η απάντηση είναι όχι. Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις τη για τι αναπτυσσόμενες χώρε ή για τι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε είναι γιγαντιαία. Αναρωτιέμαι πώς θα μεταφράσουν οι διερμηνείς αυτή τη λέξη ginormous. Είναι καταστροφικές οι επιπτώσεις για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες αλλά και για τις χώρες μεσαίων εισοδημάτων. Αυτές τιμωρούνται ό,τι και να συμβεί ε, είτε στα πακέτα βοήθειας που λαμβάνουν και είτε στα εισοδήματα που λαμβάνουν σε, καλούς, σε καλές εποχές. Η Μποτσουάνα αποτελεί ένα εξαιρετικό ε, παράδειγμα, μια χώρα μεσαίου εισοδήματος με τεράστιο πλούτο, χρησιμοποιεί τον πλούτο της προς όφελος του πληθυσμού της στο ιστορικό, ιστορικά έχει δεσμευτεί ε, με καταπληκτικά αποτελέσματα για την πρόληψη του AIDS, του AIDS, για την υγεία, για την εκπαίδευση, αλλά και για άλλα ζητήματα. Αυτή η χώρα σήμερα υποφέρει λόγω της ε, παγκοσμίας ύφεσης. Επίσης ε, έχουμε και τη συζήτηση όσον αφορά το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εμείς ε, στο Κοινοβούλιο. Έχουμε επιχειρηματολογήσει εδώ και πολύ καιρό λέγοντας, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικού τρόπους χρηματοδότησης, ενδεχομένως ε, φόρο ε, ανταλλαγής ε, τίτλων. Θα μπορούσε να προσφέρει ένα δισεκατομμύριο ο φόρος εμπορίας γεωργικών ειδών. Δηλαδή το να γίνεται ε, κέρδος, το να κερδοσκοπούν άνθρωποι είναι ηθικά απαράδεκτο σε αυτό το τομέα. Να πουλούν κάτι πολύ ακριβά το που έχουν αγοράσει για τίποτα. Ε, η χρήση των ορυκτών για να χρηματοδοτούνται οι συγκρούσεις είναι τρομερό. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να καλύψουμε αυτό το χάσμα. Ε, ώστε οι χώρες που λαμβάνουν πόρους από περιοχές ε, όπου υπάρχουν συγκρούσεις δεν θα πρέπει να μπορούν να τα πουλήσουν σε μας. Ο φόρος εξόρυξης ορυκτών για παράδειγμα είναι άλλη μια επιλογή. Θέλω λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε δημιουργική σκέψη, να χρησιμοποιήσετε δημιουργική σκέψη στην Κομισιόν. Εγώ θεωρώ σύμμαχο την Κομισιόν, φίλο μας, ε, δεν δέχομαι αυτό που συμβαίνει σε άλλες ε, επιτροπές όπου εμείς είμαστε οι καλοί και η Κομισιόν ε, είναι τα κακά παιδιά. Οι δεσμεύσεις μας πιστεύω και οι προθέσεις μας είναι ίδιες. Θέλω εμείς να βοηθήσουμε την Κομισιόν να ε, ενισχύσει την πυγμή της ώστε να διασφαλίζει ότι τα κράτη-μέλη που λαμβάνουν δεσμεύσεις θα τηρούν αυτές τις δεσμεύσεις. Διαφορετικά οι συνέπειες όταν αυτές οι χώρες ε, δεν λαμβάνουν μέρος ε, είναι σημαντικές. Η ομάδα μου θα υποστηρίξει ιδιαίτερα την πρώτη ψηφίσματος. Ε, αναμένουμε τις απαντήσεις και την απόκριση. Προς το παρόν έχουμε μία τροπολογία, διαγραφή στην παραγραφό 17, διότι οι συγκρίσεις, comparisons, πιστεύω δεν βοηθούν Θέλουμε λοιπόν να διαγράψουμε την πρόταση like the bricks. Επειδή οι συγκρίσεις τέτοιου είδους δεν βοηθούν. Υπάρχουν προβλήματα στην Ινδία τα οποία αν εμείς ε, τα προβλήματα ένδειας και λοιπούς διατροφής και έλλειψης υγείας δεν θα επιληθούν αν εμείς ε, δεν συμμετέχουμε σε αυτά. Όπως είπε μια φορά ο Όσκαρ Βάιλντ, οι συγκρίσεις είναι απέσιες. Θα πρέπει να τη διαγράψουμε λοιπόν. Εάν κάποιος ωστόσο έχει να μας κάνει μια πολύ συγκεκριμένη σύγκριση η οποία θα επιφέρει αλλαγή θα μπορέσουμε να τη λάβουμε υπόψη μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για το έργο της και να ενθαρρύνω τη συνεργασία μαζί μας ώστε οι δεσμεύσεις της ε, Κομισιόν και του Κοινοβουλίου να προωθηθούν με καλή πίστη. πρόθεσή μας είναι να τις επιτύχουμε. Δυστυχώς τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν την οικονομική κρίση ως ε, δικαιολογία, όχι αιτία, για να μην τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε καλές εποχές. Εύκολο είναι κανείς να κάνει δεσμεύσεις όταν τα πράγματα πάνε καλά. Όταν ε, οι φίλοι σου δυσκολεύονται, ε, δυσκολεύονται τότε. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρνς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεπετάξουμε μια συζήτηση εύκολα έτσι σε ό,τι αφορά την κατανομή ανεπτυξιακής βοήθειας και θα βασιστώ στο τελευταίο τμήμα της παρέμβασης του Μάικλ και θα συνεχίσω από εκεί. Δεν ε, θα μπω στην ουσία του θέματος γιατί θα μακρηγορήσω όσο αν συζητούσαμε το φύλλο των αγγέλων. Είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε μια απάντηση κατηγορηματική, αλλά για να διευκολύνουμε τη συζήτηση, στο διάλογο προς το μέλλον, θα έπρεπε την αναπτυξιακή βοήθεια που απευθύνεται κατά κύριο και πρώτο λόγο σε χώρες που πρέπει να αντιμετωπίσουν ε, την φτώχεια και να κάνουμε μία διάκριση. Έχουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά μέσα σε αυτές υπάρχουν κάποιες που δεν μπορούν καν να επιβιώσουν. Φτώχεια υπάρχει στην Ινδία, υπάρχει στην Κίνα, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά οι χώρες αυτές έχουν τα μέσα να καταπολεμήσουν τη φτώχεια. Και ουσιαστικά όχι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, αλλά ο προπολογισμό ο κρατικός των χωρών θα χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση της φτώχειας σε αυτές τις χώρες. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς λοιπόν όταν ε, παρουσιάζουμε τα πράγματα και τους λογαριασμούς. Και θα πρέπει να κάνουμε και κάποιους υπολογισμούς. Τι είναι απαραίτητο και τι δεν θα ήταν 100% απαραίτητο. Πρώτο σημείο αυτό. Και δεύτερο και τελευταίο είναι η αξιολόγηση της ε, πολιτικής της Κομισιόν από ομοτήμους. Ποιοι είναι οι ομότιμοι στην προκειμένη περίπτωση είναι το ερώτημά μου και ποιος θα είναι ο βαθμός συμμετοχής των μελών της δικής μας Επιτροπής στην άσκηση εξολόγησης από ομοτήμους στο πλαίσιο του ΟΣΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι χρήσιμο εγχείρημα. Είναι ενδιαφέρον να συμμετάσχουν ε, διάφορες επιτροπές σε αυτή την άσκηση, σε αυτό το εγχείρημα. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί κατά τη συζήτηση αυτή στον ΩΣΑ που θα γίνει παρουσία όλων των πρέσβεων του ε, ΩΣΑ όταν θα εκτεθεί ε, στις ε, ερωτήσεις η Κομισιόν αν θα μπορεί και το Κοινοβούλιο να εκπροσωπηθεί επαναλαμβάνω. Κύριε Κάσμα θέλετε κάτι να προσθέσετε. Όπως μου υπενθύμισε κάτι ο κύριος Γκούρινς θα ήθελα να το θίξω ε, συμφωνώ με την ερώτηση για τους ομοτήμους, αλλά θα ήθελα να πω ότι όταν ε, πρώτα άκουσε να μιλάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για duck peers, φαντάστηκα ότι θα μπουν ε, μεγάλες πάπιες στο κοινοβούλιο. Ducks. Μετά κατάλαβα φυσικά ότι ήταν DAC αυτό για την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας. Χαίρομαι λοιπόν που το διευκρινίσαμε αυτό. Μάλιστα. Η Κομισιόν θέλει να λάβει εκ νέου το λόγο. Νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω μόνο εν μέρη στο ερώτημά σας για το ποιο είναι οι ομότιμοι, ποιοι ε, ε, εξετάζουν την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση είναι η Ιαπωνία και η Νορβηγία. Για το δεύτερο τμήμα της ερώτησης δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν είμαι από την υπηρεσία την αρμόδια, αλλά θα διαβιβάσω το ερώτημά σας και νομίζω ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσω και αυτό με την γραμματεία την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Πριν ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών στην πρόταση ψηφίσματος 22 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα και ψηφίζουμε στις 11 Οκτωβρίου. Στα διάφορα υπάρχει κάτι. Όχι. Επομένως, επόμενες συνεδριάσεις. Η επόμενη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες 4 Οκτωβρίου 9 έως 12.30 και 3 έως 6.30. Ε, 10 Οκτωβρίου από τις 3 έως τις 6.30 και 11 Οκτωβρίου 9 με 12.30 και 3 με 6.30. Να μην ξεχάσετε την επόμενη φορά να φέρετε τις κάρτες ψηφοφορίας να είστε και στην ώρα σας και έτσι κυρίω τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής μας και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Καλή όρεξη.